Κυρίες και κύριοι, ψηφοφορίες. Έχουμε πολλά σημεία σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη. Απλουστευμένη διαδικασία. Καταρχάς έχουμε την έκθεση του κυρίου Σίμψον. Συμφωνία με την κυβέρνηση της Μογγολίας. Είναι νομαστική η ψηφοφορία και αρχίζει τώρα. Σε Πέρασε. Ψήφισαν 479, 456 υπέρ 21 κατά δύο εποχές εγκρίνεται. Επόμενο θέμα στη μέση διάταξη. Άλλη έκθεση με προσθεμένη διαδικασία πάλι του κυρίου Σίμψον. Συμφωνίες για τις αλλάσεις μεταφορές Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κίνας. Η κυβέρνηση συγκεκριμένα Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Σε Ψήφισαν 588 υπέρ 558 κατά 19 αποχές 11 εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Πάντα με την απλουστευμένη διαδικασία ακολουθεί η ψήφιση της έκθεσης του κυρίου Μπέγκε. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρασε. 610 υπέρ, 581 κατά 23 αποχές 6 εκδίδεται. Ο κύριος Σέβεριν έχει το λόγο. Ε, ε, yes, ε, I want to say that my... Θα ήθελα να σας πω ότι το μηχάνημα έχει εδώ δεν λειτουργεί. Θα σας βοηθήσουμε, αν ένα Έχω το λάθο μηχάνημα που κατάλαβα, συγγνώμη. Πάντα απλουστευμένη διαδικασία, άλλη έκθεση του κυρίου Μπέογκε. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. διατάξεις. Ψήφισαν 616, 578 υπέρ, 26 κατά, 12 αποχές εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση, πάντα με την ίδια διαδικασία, της κυρίας Χάουγκ. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, αριθμός 6 κάθετος 2009. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2009. Ονομαστική ψηφοφορία, μοναδική με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αρχίζει τώρα. Εψήφισαν 641, έλαβαν υπέρ 600, κατά 8, 33 αποχές, εγκρίνεται. Πάντα με την ίδια διαδικασία ακολουθεί η έκθεση της κυρίας Χάουκ για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 7, κάθε του 2009. Πάντα μία ψηφοφορία, ειδική πλειοψηφία, ονομαστική, που αρχίζει τώρα. Σε cierra la ε, πέρας. Ψήφισαν 642, 605 υπέρ, 23 ε, κατά, 14 αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια διαδικασία ακολουθεί η έκθεση κυρία Χάουκ το θέμα του σχέδιου διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 8 του 2009. Μία και μοναδική ε, ψηφοφορία που αρχίζει τώρα και χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. να ψήφισαν 651, 594 υπέρ, 27 κατά 30 αποχές. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνονται εδώ οι ψηφοφορίες και περνούμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Δεν έχει ζητήσει κανείς προφορική, εάν θέλετε, γραπτός. γιατί αποστείλετε στην Προεδρία. Διακόπτεται η συνεδρία σήμερα τις 11.30 όπου θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.